σκέφτηκα μόλις πριν από δύο λεπτά ότι μου ζητούν να κάνω μία ανακοίνωση για ένα πολύ τραγικό γεγονός το οποίο θέλω τώρα να σας ανακοινώσω. Με μεγάλη θλίψη και συντριβή μάθαμε σήμερα τα γεγονότα στο Βίνεντεν, στην Βάδη Βιρτεμβέργη, στην ε, Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία το ότι 15 παιδιά σκοτώθηκαν με τραγικό, 15 άνθρωποι μάλλον σκοτώθηκαν στην ε, Ρεάλ Σούλε, στο ειδικό αυτό γυμνάσιο, από ένα 17χρονο πρώην, μαθητή της σχολής, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, δύο από τους οποίους τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή αυτή πυροβολισμών. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να τονίσω την βαθιά μου συμπαράσταση και τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων. Τα θύματα ήταν αθώοι μαθητές και μαθήτριες καθώς και τρεις καθηγητές της σχολής. Αυτή η τραγωδία λαμβάνει χώρα έξι μήνες μετά από μια αντίστοιχη ενέργεια στο Κάου Αριού στην Φινλανδία και εμείς ως υπεύθυνη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό, ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε τέτοια γεγονότα να εμποδιστούν και να μην επαναληφθούν ποτέ στο μέλλον. Εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τη δική μας πλευρά. Υπάρχει ένα άλλο τραγικό γεγονός επίσης και στην Αλαμπάμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και πάλι κάποιος ο οποίος κατελήφθη από αμόκ σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους μέχρι πρωτού στρίψει το όπλο του εναντίον του εαυτού του. Θα ήθελα και πάλι εξ όλων μας, όλων σας να εκφράσω την αλληλεγγύη μας με τα θύματα και την συμπαράστασή μας προς τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να σας ζητήσω να τιμήσουμε τη μνήμη των φωνευθέντων. Ich danke Ihnen. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτήν την τραγική ανακοίνωση θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Τα χθεσινά πρακτικά έχουν ήδη μοιραστεί, υπάρχουν παρατηρήσεις από αυτόν.